Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem sich der Raum nun doch zu füllen scheint. Γεια σας. Συνάδελφοι, σιγά σιγά γεμίζει η αίθουσα. Αργά αργά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Κοιτάξτε, πρόθεσή μου είναι να βοηθήσω τους συναδέλφους που θέλουν να δουν τον αγώνα λίγο αργότερα, τουλάχιστον Ας δουν το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, εγώ θα πατήσω γκάζι και ζητώ την κατανόησή σας. Δεν θα έχουμε πολύ καστιάι και δεν θα υπάρξουν και τόσοι, πόσες πολλές συνεδριάσεις των σχεδόν γιατί πολλοί κάθονται ήδη μπροστά στην τηλεόρασή τους. Πάμε στο σημείο 1 έχετε κάποια σχόλια όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Από πλευρά διερμηνέων, θέλω να σα μιλήσουμε για την υπέρβαση του ωραρίου. Οι διερμηνεί συνεχίζουν για τέταρτη εβδομάδα τι κινητοποίησει για τι συνθήκε εργασία, καθότι η διοίκηση δεν έχει έρθει σε καμία επαφή μαζί μα για την επίλυση τη εργασιακή διένεξη. Σα πληροφορούμε ότι η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώ την προβλεπόμενη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Ω προ την ημερήσια διάταξη, έχετε παρατηρήσει ε, για τα πρακτικά. Δεν βλέπω αντιρρήσεις για το σημείο 3 της ανακοινώσεις δεν έχω και να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 4 έκθεση COFOT για την απλούστευση και την εναρμόνιση κάποιων διατάξεων και κανόνων για το ΦΠΑ και θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή μας τον Τζέπε Κόφωτ για την έκθεση του η τη συστήματο για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών. Ευχαριστώ, Πίτερ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικό, γιατί ε, πολλοί συνάδελφοι έχουν και άλλα να κάνουν σήμερα, γι' αυτό καλύτερα να ολοκληρώσουμε νωρί. Ε, ευχαριστώ για τη συνεργασία. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και μετά από σχολαστική εξέταση των τροπολογιών, ε, έχω μεγάλη αισιοδοξία γιατί έχουμε πολύ. Ε, καλή βάση για τις συμβαστικές τροπολογίες. Πολλές τροπολογίες ε, με εύστοχες ε, προσθήκες, ε, διευκρινήσεις και μνήες εμπλουτίζουν το κείμενο. Πολλές μάλιστα τροπολογίες ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση και καλύπτουν τουλάχιστον εν μέρη τα ίδια πολιτικά ουσιαστικά σημεία που καλύπτω και εγώ στην έκθεσή μου. Γι' αυτό και λοιπόν, θα ήθελα να σα προτείνω διάφορε συμβαστικέ τροπολογίε με βάση τι δικέ σα τροπολογίε Θα σα τι μοιράσω πριν την επόμενη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών. Και πριν περάσουμε σε, αυτό το, σε αυτή την κρίσιμη φάση, θα ήθελα ω αρμόδιο εισηγητής να πω λίγα λόγια για το πώ σκοπεύω να ζητήσω τη συνένεσή σα ε, για το μέλλον αυτό το θέμα. Θέλω μια ανοιχτή, αποτελεσματική και χωρί αποκλεισμού διαδικασία και για αυτό θα σταθώ σε τρία για μένα σημαντικά σημεία. Καταρχήν, δεν θα δεχτώ καμία αποδυνάμωση του κειμένου ή συρρήκνωση του πεδίου εφαρμογή του. Η έκθεση, ε, η πρόταση που έχουμε είναι ισορροπημένη μεταξύ της πραγματικής και επιτακτικής ανάγκης διευκρίνηση και απλούστευσης του διασυνοριακού ΦΠΑ και της ε, κρίσιμης ανάγκης για αποτελεσματικές εναρμονισμένες ασφαλιστικές δικλείδες για να αποτρέψουμε την απάτη στο ΦΠΑ. Αυτά τα δύο βασικά τμήματα ε, του πακέτου είναι απολύτως απαραίτητα. Επίσης, θέλω να κρατήσουμε αμετάβλητα το πεδίο εφαρμογή του κειμένου. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι μπορούμε ε, θα έπρεπε να αντισταθμίσουμε προσωρινές λύσεις εξαιρέσεις ή ειδικού κανόνες. Επίσης, ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε όσον νούπο σε συμφωνία και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να την προλυάνω και να την διευκολύνω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Γέπε για δύο λεπτά. Ε, το λόγο έχουν οι σκιοδησηγητές. πρώτη κυρία Ιβάνα Μάλετης εκ μέρους του ΕΛΚ. Ε, μάλλον όχι. Ο, ο αναπληρωτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε το Γέπε Κόφωτ για την σύντομη εισαγωγή. Η Ιβάνα Μάλετης μου ζήτησε να την αντικαταστήσω σήμερα για την ισκιώδη συγκήτρια στο θέμα αυτό, στην έκθεση αυτή. Η προσωρινή λύση για το σύστημα ΦΠΑ για τις διασυνοριακές συναλλαγές υιοθετήθηκε πριν από 25 χρόνια και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι προσωρινές λύσεις γίνονται μόνιμες, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Οι σημερινές αλλαγές είναι κάποιες γρήγορες προσωρινές λύσεις, μαγικές λύσεις των προηγούμενων προσωρινών λύσεων εν ώψη ενός προσωριστικού συστήματος ε, με βάση την αρχή του προορισμού για τη φορολογία ΦΠΑ. Με τις αλλαγές αυτές έχουμε τη νέα έννοια του πιστοποιημένου υποκειμένου στο φόρο και μάλιστα δεν ξέρω αν έχει νόημα να το κάνουμε τώρα με ένα quick fix, με μια σύντομη μαγική λύση ή να το αφήσουμε για αργότερα προκειμένου να παραμείνει στο οριστικό σύστημα ΦΠΑ. Αν μπει τώρα αυτή η πρόταση των πιστοποιημένων ε, υποκειμένων στο φόρο, η Ιβάνα Μάλετη συμφωνεί με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω και να αποσαφηνίσουμε την έννοια και τα κριτήρια του πιστοποιημένου υποκειμένου στο φόρο ε, με εκτελεστικούς κανονισμούς και ε, εξονυχιστικές και δελεχείς καταθεντήριες γραμμές. Μάλιστα, ε, το One Stop Shop, η μονοαπευθυντική θηρίδα, είναι ο πυρήνας του συστήματος, του οριστικού συστήματος με βάση την αρχή προορισμού, χωρίς επιπλέον όμως επιβαρύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό, για να ε, ετοιμάσουμε αυτό το σύστημα, ε, θα πρέπει να παρατείνουμε τη, τη μονοπευθυντική θηρίδα για να καλύψουμε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ε, γίνονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση το παρόν σύστημα. Επίσης, η κυρία Μάλα θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε και ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών ΦΠΑ. Και στην αρχή μπορεί να είναι online πλατφόρμα, ώστε να μπορέσουν τα κρατημέρια να διευθετούν τις διαφορές τους, κάτι που η άλλη, όταν η άλλη διαδικασία δεν αποφέρει καρπούς. Ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάποιες προσεγγίσεις ε, για να αυληθούν οι διαφορές και θα προβλέπει και διαδικασίες για τη διαθέτηση των διαφορών. Μία πλατφόρμα επίλυσης διαφορών θα πρέπει να είναι προσβάσιμη, εύχρηστη και με χρονικά περιθώρια για την επίλυση των διαφορών. Εν κατακλείδη, η Ιβάνα Μάλετιτς τονίζει ότι η δημιουργία ε, ενό ενιαίου χώρου ΦΠΑ είναι απαραίτητη για να μειωθεί το κόστο συμμόρφωση για τι επιχειρήσει, να μειωθεί ο κίνδυνο τη διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ και γενικώ για να απλουστεύσουμε τι ε, διαδικασίε που αφορούν το ΦΠΑ. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα ενισχύσει την αγορά και θα δημιουργήσει καλύτερε προποθέσει για το διασυνοριακό εμπόριο. Κάτι άλλο που θα πρέπει να περιλαμβάνουμε σε αυτά τα quick fixes που προτείνονται, σε αυτέ τι σύντομε μαγικέ λύσει, είναι τι προσωρινέ λύσει, είναι να ληφθούν υπόψη τεχνολογικέ εξελίξει, η ψηφιοποίηση και αλλαγή στα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώ και να ληφθεί υπόψη και η παγκοσμιοποίηση τη οικονομία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ Μπέρκαρτ κύριε Ζούνε από το ECR, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Γέπε. Όλοι συμφωνούμε. Χρειάζεται εξυγχρονισμό στο ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ, να μειωθεί το διοικητικό άκθο, να καταπολεθεί μια απάτη στο ΦΠΑ. Χάρηκα από αυτά που είπε. Χρειάζεται γρήγορη συμφωνία. Συμφωνώ. Απόλυτα κι εγώ. Για το γενικότερο θέμα θέλω να μιλήσω και μετά για τι γρήγορε λύσει. Καταλαβαίνω τη λογική. Ε, η αρχή με βάση τον προορισμό είναι καλή αρχή. Θέλουμε να δούμε ποιο θα είναι ο αντίκτυπο στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αν θα αυξηθεί το διοικητικό άχθο κλπ. Γι' αυτό έχουμε σχετικέ τροπολογίε. Βασικό ερώτημα και θέμα δεν είναι ότι παρακολουθούμε τη λογική που ακολουθούμε, αλλά θέλουμε να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί, αλλά και ποιε θα είναι οι νομικέ επιπλοκές, εάν είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Και όπως είπες, θα εξετάσουμε το πεδίο εφαρμογή ή όχι. Γι' αυτό υποβάλαμε σχετικέ τροπολογίε. Είχαμε τροπολογίε για περιορισμό του πεδίου εφαρμογή. Θα θέλαμε να αποφύγουμε νομικέ επιπλοκέ, καθυστέρηση εφαρμογή των γρήγορων ε, λύσεων, των quick fixes. Αυτή είναι η προτεραιότητα τα μέτρα αυτά τα διευθυντικά να εφαρμοστούν ταχύτερο δυνατόν. Και γι' αυτό εστιαζόμεθα σε αυτό το σημείο κυρίως της τροπολογίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάντερ για την Άλντε. Τέρι Κόνλι δεν είναι εδώ. Άλλος που θέλει να μιλήσει. Όχι. Εκ μέρους του. Όχι. Εν τη αυτή περίπτωση. Μόλις... Για τους πρασίνους. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Υποστηρίζουμε την πρόταση. Είπαν και άλλοι συνάδελφοι ότι απλουστεύεται το σύστημα του ΦΠΑ και καταπολεμούμε την απάτη και απομακρυνόμαστε το περίπλοκο προσωρινό σύστημα και πάμε προς ένα μόνιμο σύστημα. Ο πιστοποιημένο φορολογούμενος αυτό το σύστημα, δημιουργεί εμπιστοσύνη για τι επιχειρήσει, όπου σε δυσυνορικές πωλήσει θα πληρώνει επιχείρηση χώρα προορισμού το ΦΠΑ. Θεωρούμε ότι είναι καλή πρόταση αυτή. Απλουστεύει την κατάσταση κυρίως για αυτούς που αναγνωρίζονται ως ε, φορολογούμενα ε, πρόσωπα. Εμείς που έχουμε ασχοληθεί με τη φοροαποφυγή σε διάφορες επιτροπές όσον αφορά το ΦΠΑ, ξέρουμε ότι πάντα όταν προσπαθούμε να βρούμε λύσεις υπάρχουν κενά και νομοθέτε πρέπει να είναι προσεκτικοί. Υποστηρίζουμε την ένα του πιστοποιημένου φορολογούμενου καταρχήν, αλλά οι τροπολογίε 43, 47 και 51 εστιάζονται επί αυστηροτέρων συνθήκων υπό τις οποίες αποκτά αυτό το καθεστώς με επιχείρηση. Μία από τις καλύπτει την περίπτωση ιστορικού εγκληματικών αδικημάτων που ένας λόγος να εξαιρεθεί κάποιο από τον τύχη αυτού του καθεστώτος ή αδικήματο σχετίζονται με οικονομική δραστηριότητα του ετούντος ε, και αρκετά άλλα. Πρέπει λοιπόν να ισχύουν οι κατάλληλε συνθήκε, ούτω ώστε να μην μπορεί κανεί να κάνει ε, ψευδεί αιτήσει και να θεωρείται φορολογούμενο και να μην πληρώνει τα ποσά που θα έπρεπε. Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνεδρίαση των σκιωδών την επόμενη εβδομάδα και σίγουρα θα βρεθεί κάποια ε, συμβαστική λύση, κάποιες συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Μόλι, για την ΚΟΕ. Μιλάει εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος, δεν τον ακούνε οι διερμηνείς, δυστυχώς. Η ε, Μπάρμπαρα Κάπελ θα έπρεπε να είναι εδώ, δεν είναι. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, Γκουε, κυρία Παπαδημούλη και μετά η ΕΝΕΦ, η κυρία Κάπελ. Αλλά κανείς από τους συναδέλφους δεν είναι εδώ, σε αυτή τη φάση, οπότε πάμε πίσω στον εισηγητή, στο Γέπε Κόφορντ. Ευχαριστώ. Όπως προανέφερα, θα επεξεργαστούμε σχέδιο συμβιβαστικού κειμένου. Θα συνεδριάσουν σκιώδες την επόμενη εβδομάδα και με τα σχόλιά σα, που ήταν θετικά σίγουρα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου σε μια λύση η οποία θα είναι καλή και ταχεία και αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω κάτι ότι στις 3 Σεπτεμβρίου στην Οίκον και στην Ολομέλεια πιθανότατα στην πρώτη σύνοδο του Οκτωβρίου. Ε, λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε, να πάμε στο σημείο 5 της ημερησίας σας. Ε, τροποποίηση της 2612 ε, όσον αφορά το προστιθέμενο, τη στάθμιση του προστιθέμενου αξία του ΦΠΑ. Ο κ. Τζάνι για, το, για τους σοσιαλιστές είναι Λοιπόν, ο Τίμπορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ Πίτερ. Καταρχάς, Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητές για την επικοδομητική του στάση και την εργασία τους. Έχουμε 52 τροπολογίες από διάφορες πολιτικές ομάδες. Κοινή προσέγγιση. Αυτό φαίνεται από τις λίγες σχετικές τροπολογίες που υπευλήθησαν και διότι το περιεχόμενο των τροπολογιών δεν αποκλίνει πολύ. Την περασμένη εβδομάδα έγινε η πρώτη συνεδρία των σκιωδών Εκεί συζητήσαμε 11 ενδεχόμενες συμβαστικές και με τα χαράς ανακοινώνω ότι έχουμε βρει την κατάλληλη πλειοψηφία σχετικά με όλα τα κρέμοντα ζητήματα. Από ό,τι γνωρίζω, οι εκπρόσωποι των περισσότερων κομμάτων ήδη συμφωνούν επί της βασικής γραμμής. Δηλαδή πράγματι υπάρχει ανάγκη να αντικατασταθεί το παρόν μεταβατικό σύστημα και να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρατών μελών. Επίσης συμφωνούμε επί της ανάγκης να τεθεί τέρμα στον κατακαιρματισμό των άχρηστο του συστήματος του ΦΠΑ που δημιουργεί εμπόδιο για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Δεν έχουμε μεγάλες διαφωνίες ούτε επί της προτάσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το τελικό σύστημα του ΦΠΑ για τη φορολόγηση εμπορίου μεταξύ κρατών μελών θα εδράζεται επί της αρχής της φορολογήσεως στο κράτος μέλος προορισμού φαίνεται ότι οι πολιτικέ ομάδε συμφωνούν με εναρμονισμένου κανόνε που θα είναι λιγότερο περιοριστικοί και έτσι τα κράτη-μέλη πέρα του να εφαρμόσουν ένα, ένα ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 0%. Σύμφωνα με την πρόταση, παράρτημα 3 αντικαθίσταται απαρνητικό κατάλογο που θα αναφέρει σε ποια αγαθά ή υπηρεσίε δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα μειωμένα ποσοστά. Όμω δεν υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά την αλλαγή. Κάποιε τροπολογίε επίση υπευλήθησαν για μια συμπληρωματική λίστα θετική. Θεωρώ ότι τα μειωμένα ποσοστά και εξαιρέσεις θα αφαιρούν τον τελικό καταναλωτή και πρέπει να δοθεί κατάλληλη προτεραιότητα. Να αφορά αγαθά υπηρεσίε που έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ω συζητητή και μέλο ομάδα σοσιαλιστών, απευθύνω έκκληση προ τα κράτη-μέλη να αποφύγουν την χρήση ε, ε, για ε, κάποιων ποσοστών για τα είδη πολυτελείας, μειωμένων ποσοστών. Για να ευκολύνουμε το εμπόριο στην ενιαία αγορά και να καλύψουμε τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προτείνουμε να υπάρχει ένα, μια πύλη στο διαδίκτυο για το ΦΠΑ γιατί στην Ευρώπη για να δίνει γρήγορα πληροφορίες επιχειρήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ στα διάφορα κράτη-μέλη. Επ' αυτού να ευχαριστήσω εκ νέου τους και ηγητές και τους άλλους συναδέλφους ευρωβουλευτές που εργάστηκαν με αφοσίωση και αυτό βοήθησε να βελτιώσουμε το σημαντικό το αυτό εργαλείο. Συνεχίζοντας με την υποστήριξή σας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία που δείξατε μέχρι τώρα για την επιτυχή βελτίωση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τιμπορ. Λοιπόν, ο Βέρνερ Λάγκεν για το ΕΛΚ. Να του δώσουμε το λόγο αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν είναι έκτακτη συνεδρίαση αυτή. Είναι μια συνεδρίαση που είχε κοινοποιηθεί, είχατε ειδοποιηθεί. Δεν είχαμε όμως τότε το πρόγραμμα αυτό, το, δεν ξέραμε και το πρόγραμμα αυτό του, των ποδοσφαιρικών αγώνων και δεν ήξερα ποιο θα προεδρεύσει. Γι' αυτό έφτασα και καθυστερημένος Και είχαν πάρει συνάδελφοι το λόγο. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Γκουαλτιέρη συνήθω έρχεται πιο αργά και το είχα συνηθίσει. Λυπάμαι λοιπόν που ήρθα και εγώ αργά. Αυτά είναι είδη εισαγωγή. Λοιπόν, πήραμε την έκθεση, είχαμε τη δυνατότητα να τη συζητήσουμε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι βλέποντας τι έχει ήδη επιτευχθεί. Υπάρχει ε, μία σειρά συμβιβαστικών λύσεων που έχουν υποβληθεί και αυτές οι συμβαστικές συνετάχθησαν βάσει των τροπολογιών που είχαν υποβληθεί. Σε αυτές οι συμβαστικές λύσεις βασικά αναφέρεται το πώς μπορούμε να καταλήξουμε με μια λογική πρόταση, σε μια λογική πρόταση την οποία το Συμβούλιο να μπορεί να την αποδεχτεί και να μπορεί να υποβληθεί και στην Ολομέλεια. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο, άρα έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε τις συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή για όλη την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Δεν έχουμε κάποια μεγάλα προβλήματα. Ε, η έκθεση αυτή δεν μας δημιουργεί πολλά προβλήματα. Πρέπει να ψηφιστεί με ομοφωνία στο Συμβούλιο και αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία, παρουσιάζουμε σαν κοινοβούλιο κάποιες προτάσεις στο Συμβούλιο. Αυτό το κάναμε και πριν τεθεί σε εφαρμογή ε, η συνθήκη της Λισαβόνας. Το ΕΛΚ αισθάνεται και θεωρεί ότι οι προτάσεις αυτές και το θέμα που συζητούμε, δηλαδή τα μειωμένα ποσοστό ο αριθμός των περιπτώσεων για εφαρμογή μειωμένων ποσοστών πρέπει να ε, μειωθεί. Έχουμε πολλές εξαιρέσεις αφορά το επίπεδο ΦΠΑ λόγω πολλών μέτρων που είχαν θεσπιστεί το, τη δεκαετία των 90 και συνεχίστηκαν. Όλα αυτά τα ειδικά καθεστώτα. Ένα από τα πράγματα που θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν είναι να αποφασίζουμε επί πραγμάτων που σε άλλες εκθέσεις όπως το e-books ε, έχουν αποφασιστεί. Ε, ίσως είναι ενδεδειγμένο να κάνουμε κάποια αμνία στη τηλεολογική σκέψη, αλλά όχι στο διατακτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια αρνητική, έναν αρνητικό κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών. Για αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες δεν μπορούν να υπάρξουν μειώσεις ποσοστών ΦΠΑ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι θετικό, αλλά πρέπει να επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια αυτός ο κατάλογος, να επικαιροποιείται, να ενημερώνεται τακτικά και όλες οι ομάδες συμφωνούν ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε την κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι θα πρέπει να δίδουμε καλύτερες πληροφορίες στους καταναλωτές. Να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα ενημέρωση για να μπορούν εύκολα να ενημερώνονται οι καταναλωτέ για τα διάφορα ποσοστά ΦΠΑ. Υπάρχει μια τροπολογία των πρασίνων για την οποία έχω κάποιε αμφιβολίε. Δηλαδή, πέρα από την ιδέα των μειωμένων ποσοστών ΦΠΑ έχουμε και πολύ πολύ μειωμένα ποσοστά που είναι πιο χαμηλά το 5% και υπάρχουν κάποια παραδείγματα από διάφορες χώρες και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Χρειάζεται συζήτηση πραγματικά. Εν τω μεταξύ το Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει το χαμηλότερο ποσοστό το 15%. Υπήρχαν πάντα, πάντοτε κενά ε, το καθεστώς ίσχυε για πενταετία και ο εισηγητής προτείνει ένα νότατο όριο 25% και θυμάμαι ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο προσπαθήσαμε εδώ και 15 χρόνια άνευ επιτυχία. Το Συμβούλιο απέρριψε αυτή την ιδέα τότε. Λοιπόν, σκεφτείτε το. Υπάρχει μόνο μία χώρα που έχει ένα ποσοστό που είναι πάνω από 22% και είναι η Ουγγαρία αυτή. Εκεί έχουν 27%. Είναι η χώρα του συγητή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για την μείωση αυτού, αλλά πραγματικά μόνο μια χώρα θα πληγεί από κάτι τέτοιο, θα επηρεαστεί από κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία και αρκετά εύκολα και να υποβάλουμε και κάποιες συστάσεις για τις 3 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος πάλι για τους και φινδαρισμιστές. Α, μόλις έφυγε από την αίθουσα. Από την δεν θα πάρει κάποιος στο λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για την κατεύθυνση που έχει πάρει αυτή η έκθεση. Γι' αυτό και έχουμε καταθέσει τροπολογίες. Θα ήθελα να βελτιώσουμε την ομολογία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την, την ομοθεσία συγγνώμη, αποφεύγοντας επιβαρύσεις και επίσης να πλουστεύσουμε το σύστημα ΦΠΑ για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Βέβαια, ε, φαίνεται ότι γίνεται ένας πληροδοτικός διαγωνισμός που θα προσφέρει περισσότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να ε, πριδανεύει η κοινή λογική και μερικές φορές ε, επεμβαίνοντας σε συστήματα ΦΠΑ των κρατών μελών. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση για επάνωδο στην κοινή λογική. Εμείς με τις τροπολογίες μας θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μηχανισμούς ε, σωστής παρακολούθησης. Ε, και γι' αυτό έχουν, θα συμφωνήσουμε με κάποιες τροπολογίες συναδέλφων, αλλά μερικές τροπολογίες των σιωλιστών και των πρασίνων είναι περιτές. Και δεν νομίζω ότι θα βελτιώσουν τη φορές πρακτική ικανότητα των κρατών μελών. Επίσης, ε, ε, με τα 2 εκατομμύρια ευρώ που προτείνεται ως κατόφλι δίνεται η δυνατότητα για πολλές ε, φορολογικές καταχρήσεις. Επίσης θα ήθελα να δεχτείτε ε, τις τροπολογίες μας ε, για το άρθρο 274C, για τον τρόπο τιμολόγησης. Γιατί οι πλουστεύσεις που προτείνεται είναι υπερβολικές. Και το τιμολόγιο είναι μια απόδειξη πληρωμής και είναι απαραίτητο στοιχείο. Το ECR δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις τροπολογίες του εισηγητού που ανεβάζει το κατόφλι από τα 2 στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί ήδη για τα 2 εκατομμύρια ευρώ έχουν πολλά κρατημέλη πρόβλημα. Το θεωρούν υπερβολικά υψηλό κατόφλι. Και θα ευνοήσει περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, ε, για την οριστική προθεσμία σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή ε, του ψηφίσματος. Εγώ θα ήθελα να έχουμε τις συντομότερες δυνατές προθεσμίες. Επίσης, είναι περίπλοκο αυτό το θέμα και συμβαδίζει με άλλα, άλλες προτάσεις φορολογικές, αλλά η συνάφεια δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μπορέσουν όλο το πακέτο να, να το εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να αποφασίσουμε αν θα εγκρίνουμε την ε, πρόταση του κυρίου Σάνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κ. Ζουκ. Θα καταγράψω όσα μόλις μας είπατε για να τα πούμε και στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, γιατί νομίζω ότι ε, βιαστήκατε και μιλούσατε για το 6, κυρία Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώ να καταγραφεί ότι και εγώ ενδιαφέρομαι για το ποδόσφαιρο, παρόλο που είμαι γυναίκα μέλο τη επιτροπής αυτή. Ε, Βεβαίω με ενδιαφέρει πιο πολύ άλλο μάτσα το σημερινό. σε λίγο θα πρέπει να πάω στη Λίμπε και να πω γρήγορα πριν σχολιάσω ότι εκ μέρους του κυρίου Φάντεν Καντελάρε θα σας διαβάσω τα εξή. Χαίρομαι που η Επιτροπή έχει προτείνει τα 85.000 ευρώ ως μέγιστο όριο, σημαντικό για τις μικρές επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για τα ποσοστά ΦΠΑ, του συντελεστέ ΦΠΑ, είχαμε καλή συνεννόηση στην συνεδρία των σχεδόν την περασμένη εβδομάδα. Δεν συμφωνήσαμε στι συμβαστικέ απαραίτητε, αλλά τα πήγαμε καλά μεταξύ μα. Ήδη σημαντικό. Και συμφωνήσαμε για κατά τμήματα ψηφοφορίε σε κάποιε ειδικέ βασικέ ψηφοφορίε, όπω την 38, τη δυνατότητα των κρατών μελών να μειώσουν το συντελεστή, αν θέλουν. Αυτό νομίζω ανέφερε και ο κύριο Λάγκεν και δεν του αρέσει και πολύ. Εμεί προτείναμε δύο συντελεστέ, 10% και 5%. Η λογική μας εδώ είναι ότι η απλούστευση των συντελεστών θα διευκολύνει τις επιχειρησιακές συναλλαγές διασυνοριακά, διότι οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν πρώτα αν είναι επιλέξιμο για μειωμένο συντελεστή, 5 ή 10% επιχειρήσεις, αντί να περιμένουν να πάνε πρώτα τα προϊόντα στη χώρα και να ορίσουν του διαφορετικού συντελεστέ. Επίση, σημαντική για μα είναι η Επιτροπολογία 54. Την κλίδα ασφαλεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην είναι πάρα πολλά τα προϊόντα με μειωμένο συντελεστή. Εμείς ε, προτείνουμε ένα σταθμισμένο μεσόωρο ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή όλα τα κράτη-μέλη, το 15%. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιλέγουν λοιπόν προσεκτικότερα ποια ε, προϊόντα θα ευνοούνται από τον μειωμένο συντελεστή, όπως αυτά που έχουν ήδη χαμηλό γενικό συντελεστή, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα ας πούμε. Θα ήθελα λοιπόν οι συνάδελφοι να διαβάσουν προσεκτικά τι τροπολογίε μας, είναι σημαντικέ. Äh, Ευχαριστώ, ε, Μόλι. Για την ΚΟΕ δεν είναι εδώ ο κύριος Βιέγκας. Δεν θα πάρει κάποιος άλλος το λόγο στη θέση του. Ο κύριος Σάνι έχει πάλι το λόγο. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος θέλει το λόγο στο Κατσιάι. Όχι. Τίμπορ. Ευχαριστώ, Πέτερ. Νομίζω τα έχουμε συζητήσει διεξοδικώς στις συναντήσεις μας. Και απλώς να επαναλάβω ότι το θέμα εδώ είναι η γενικότερη αντίληψή μας για το τι είναι λογικό και τι όχι. Νομίζω ότι αυτά που συμφωνήσαμε, και αυτό είναι το σημαντικό, μας φέρνει να ξεφύγουμε λίγο από το αυστηρό πλαίσιο των εγκεφάλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και να μην ε, περιορίσουμε τα κράτη-μέλη στο τι συντελεστή θα εφαρμόζουν, βέβαια πάντοτε εντός κάποιων συγκεκριμένων πλαισίων. Εδώ θέλαμε απόλυτη σαφήνεια, όχι απλώς σαφήνεια για τα κράτη-μέλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις και ειδικώς για τις μικρομεσαίες. Νομίζω ότι η βασική καινοτομία της εκθεσής μας είναι το πόρταλ στο διαδίκτυο για τις πληροφορίες περί ΦΠΑ. Αυτό είναι κάτι που ε, το έχει στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το προωθεί στις γενικές του συζητήσεις και είναι και κάτι που θα είναι ευπρόσδεκτο από το ευρύ κοινό. Πρέπει να πω επίσης από την πλευρά του ΕΛΚ ότι η δική μας πρόταση για ενότατο όριο στον συντελεστή ΦΠΑ στο 25% θα δημιουργήσει κάποιο είδους ανάγχωμα για αυτούς που έχουν ε, πολύ μεγάλες ορέξεις και θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια. Σε κάθε περίπτωση έχουμε λάβει όλες τις συνεισφορές, δεν υπάρχουν ε, οξύς αντιπαραθέσεις, σοβαρές ε, διαφωνίες. Και ελπίζω ότι σε αυτό το αρμονικό πνεύμα θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ε, έκθεση με μια καλή συνεννόηση. Ευχαριστούμε, Τίμπορ. 3 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και θα το δούμε στην, ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Σημείο 6. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και ειδικά μέτρα για τις μικρές επιχειρήσεις. Εισηγητής ο κύριος Φάντεν Κέντελάρε. Τόμ, ευχαριστώ πρόεδρε. Παίζει το Βέλγιο απόψε. Πρέπει να είμαι τάχιστος. Να ευχαριστήσω τους κοιόδης ε, συναδέλφους για τις συζητήσει που είχαμε στην πρώτη συνεδρίαση. Και από τις τροπολογίες βλέπουμε ότι αυτό που πάνω απ' όλα επιδιώκουμε είναι η απλούσταυση. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε καλές συμβαστικές λύσεις και να ψηφίσουμε για αυτά την επόμενη εβδομάδα. Πρόεδρος, δεν υπάρχει γαλλική διερμηνία. Α, υπάρχει. Ε, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις για τις εξαιρέσεις του από το ΦΠΑ που θα αφορούν τις, τις μικρές επιχειρήσεις και δυνατότητα να τις ε, καταχωρήσουμε αυτές τις ε, επιχειρήσεις για να υποβάλουν εκθέσεις. Να δηλώνουν ΦΠΑ. Ελπίζω ότι θα προβλέψουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να το, καταφέρουν, για να το οργανώσουν αυτό τα κρατημέλη και να ζητούν τις δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά με τρόπο απλουστευμένο. Θέλουμε λοιπόν να τα απλουστευμένα δεδομένα. Η προτροπή μου λοιπόν είναι σαφή. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και αυτό για δύο λόγου. Πρώτα απ' όλα για την επιγραμμική πώληση προϊόντων και αγαθών που έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ από την διαρκή ψηφιοποίηση. Έχουμε ξεπεράσει πλέον. Ε, είναι απαρχαιωμένοι οι κανόνε περί ΦΠΑ. Αν παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τι διαδικτυακέ πωλήσει ΦΠΑ, ε, υπάρχουν πωλήσει ε, που απαιτούν να επιβληθεί δήλωση σε πέντε διαφορετικέ γλώσσε. Αυτό είναι πρόβλημα για τι μικρέ επιχειρήσει. Πρέπει λοιπόν να αποστείλουμε ένα σαφέ μήνυμα. Θέλουμε οι επιχειρήσει να αποφεληθούν από την ψηφιοποίηση και τι διαδικτυακέ πωλήσει και οι μικρομεσαίες εδώ έχουν σημαντικότερο ρόλο να διαδραματίσουν για να απαντήσουν, να, να αποκριθούν, ανταποκριθούν στις απαιτήσει του ΦΠΑ. Οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονται 0,15% ε, να διαθέσουν για να καλύψουν το πρόβλημα των δηλώσεων των ΦΠΑ. Ενώ μια μικρή επιχείρηση με λιγότερου από 20 εργαζομένου θα πρέπει να προβλέψει 0,40%. Ε, πολύ περισσότερο από ότι μια μεγάλη επιχείρηση. Πρέπει λοιπόν να τους διευκολύνουμε. Περιμένω να ακούσω τη συνέχεια των συζητήσεων και να δω ότι οι προπολογίες θα υποβληθούν ξεχωριστά. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Σάντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βασικά, εδώ δεν έχουμε πρόβλημα ιδεολογικό. Το θέμα είναι πού θα, ε, βρούμε, που θα θέσουμε τα όρια, τα ανώτατα, ανώτατα και τα κατώτατα. Θέλουμε μικρομεσαίε να είναι πιο ανταγωνιστικέ, αλλά θέλουμε να καλύπτουμε, να καλύπτουμε και το κόστο του ΦΠΑ. Άρα το θέμα είναι κάπω να διαλέξουμε ιδεολογικά, όχι πραγματικά να βρούμε συμβαστικέ λύσει. Το θέμα είναι να μα πει το ΕΛΚ ποιο νομίζω ότι είναι το καλύτερο όριο, ε, ανώτατο και κατώτατο. Η πρόταση είναι τεχνικός καλή, ε, τη την όλη διαδικασία τη στηρίζουμε. διότι επικεντρώνονται στο να μπορέσουν και οι μικρομεσαίες να συμμετέχουν περισσότερο στις διασυνοριακέ εμποροπολισίε. Ε, θα πρέπει λοιπόν εδώ Ε, εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε να μην ανοίξουμε το δρόμο για φοροδιαφυγή, ε, παραβιάσεις των κανόνων και άλλα ανεπιθύμητα φαινόμενα. Οι τροπολογίες επιτρέπουν σε κάτι μέλη που θέλουν να είναι αυστηρότερα να το κάνουν αυτό. Και σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων. Mm. Και αυτό πρέπει να το επιτρέψουμε γιατί σε, κάποιες, ε, σε κάποια κρατή πολύ μικρέ επιχειρήσει έχουν άλλη ε, βαρύτητα και σημασία από ότι για κάποιου άλλου. Η δική μου πρόταση είναι να παραμείνουμε στην αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντω. Συζητήσαμε και με προσώπου των επιχειρήσεων, με μεγάλου ομίλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρκετή πείρα στον χώρο αυτό. Εγώ θα έλεγα λοιπόν το καλύτερο είναι να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια αντίρρηση που έχω να προβάλλω ε, και θα ήθελα να την ακούσει ο εισηγητής είναι ότι τα κατώτατα όρια, αυτό που προτείνεται των 15.000 ευρώ, δεν είναι καλή ιδέα διότι στη φορολογική εξίσωση το κατώτατο όριο δυσκολεύει το, την, το, το να εξισορροπήσουν τα πράγματα μικρές επιχειρήσεις. Επίσης για τις εταιρείε με 4 εκατομμύρια κύκλο εργασιών. Αυτό μου φαίνεται λίγο υπεραισιόδοξο από κάθε προοπτική. Και μια άλλη τροπολογία που προτείναμε, η 41 να έχουν διετία αντί για ένα έτος οι μικρές επιχειρήσεις ως μεταβατική περίοδο. Γιατί εκεί που υπάρχει δυνατότητα να προβλέψουν το πώς θα πάνε τα πράγματα. Ε, την μια χρονιά μπορεί να είναι στο πάνω μέρος της καμπύλης και την άλλη στο πιο χαμηλό. Οπότε είναι καλό να έχουν δύο χρόνια για να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Αλλά αυτό μπορεί να το αποφασίσουμε και βάσει των εμπειριών που έχουν ε, οι βουλευτές και από όσα μαθαίνουν από τις εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Από το ECR ο κύριος Σόσοκ ήδη έκανε γνωστή τη θέση του, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην εκπρόσωπο των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Γενικώ ε, συμφωνούμε με την άγουσα που ακολουθεί ο Τόμ ε, και μάλιστα είχαμε μια πολύ αποδοτική και καρποφόρα συνεδρία των σχεδόν εισηγητών πριν από δύο εβδομάδες. Ε, η έκθεση, το σχέδιο έκθεση στηρίζει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η επέκταση της απαλλαγής ΦΠΑ και για τις αδοκινοτικές συναλλαγές ενισχύει την ενιαία αγορά και επίσης δίνει ενάψματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για διασυνοριακές συναλλαγές και εμπόριο. Επίσης ε, ζητά περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που επίσης είναι ε, κρίσιμο θέμα αν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ανάγκη της ενίσχυσης της ενίας αγοράς. Επίσης θέλουμε καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων αυτών και θέλουμε να συνταχθεί μελέτη επιπτώσεων για το πώς εφαρμόζεται η μονοπευθυντική θηρίδα και τι ωφέλη έχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, αν η διαδικασία πλούστευσης θα ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα, τις αρμόδιες αρχές. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε μελέτη επιπτώσεων για, για αυτά τα θέματα πριν δούμε αν είναι εφικτή μόνο, μονοπευθυντική θηρίδα. Γιατί υπάρχει ε, υπάρχουν τόσο μεγάλε διαφορέ στι επιστροφέ ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών. Για να μην αναφέρω του γλωσσικού φραγμού, ε, τα θέματα επικοινωνία και ούτω καθεξή που ανέφερε ο Τόμ. Φαίνεται ότι αρκετέ πολιτικέ ομάδε είναι υπέρ τη πρώτη. Φάνηκε αυτό στου και ηγητέ. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το σχετικό νομοθετημά καλό θα ήταν να εγκριθεί από το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κέριο ρόλο και για την ανάπτυξη αλλά και για την ευημερία. Μάλιστα. Ε, δεν βλέπω στην αίθουσα πια τον πρόσωπο των Πρασίνων, κυρία Βερμέχο από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθειά του και την, το σχέδιο έκθεσής του. Κατά τη γνώμη μας το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία και δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Γιατί όλοι ενδιαφερόμαστε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που επηρεάζονται ιδιαίτερως από την οικονομική κρίση και από την αφιλελεύθερη ε, διαχείριση που έγινε της κρίσης. Οι τροπολογίες μας ε, προσπαθούν να δώσουν λύση σε διάφορα προβλήματα, να διευκολύνουμε την οικονομική και διοικητική πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να τους προσφέρουμε τεχνικά μέσα ώστε να διευκολύνουν την οικονομική τους δραστηριότητα και απλουστεύουμε τα, τις ε, νομοθετικές διατάξεις. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια σε κάποια επιμέρους ζητήματα που για μας είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, θα πρέπει η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να μην αποδυναμώσει πλήρως τα γενικά μέτρα. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε οι μεγάλες επιχειρήσεις να μην χρησιμοποιούν τους πόρου αυτού ε, για να προσπορίζονται ίδια κέρδο θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της παράδοσης των αγαθών και της παροχής των υπηρεσιών. Κατά τη γνώμη μου, οι προτάσεις αυτές ε, προσφέρουν ασφάλεια δικαίου και καθιστούν πιο ξεκάθαρη και διαφανή τη διαδικασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και από αυτή την άποψη θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τον γιατί να κάνει μια ίστατη προσπάθεια και να δεχθεί και τις δικές μας τροπολογίες για τα σημεία αυτά. Γιατί πρόκειται για μια έκθεση που θα μπορούσε να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία και γι' αυτό αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα πλέον βήμα και μία πλέον προσπάθεια για να την εξασφαλίσουμε αυτή την συντριπτική πλειοψηφία. Ευχαριστούμε κυρία Παλώμα Βερμέχο. Άλλος κανείς παρακαλώ θέλει το λόγο. Όχι. Οπότε ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Βαντέν Κέντελαρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω ούτε κι εγώ άλλες παρατηρήσεις. ευχαριστώ. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο και πάλι. Μία μικρή παρατηρήση. Το σημείο 6 θα ψηφιστεί στην Επιτροπή στις 11 Ιουλίου και θα πάει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου η έκθεση του κ. Βαντεκέντελαρε. Περάμε στο σημείο 7. Τις οικονομικές πολιτικές ε, της ζώνης του ευρώ. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση του κυρίου Μπαγιέ, ο οποίος ε, θα μας το παρουσιάσει. Η κυρία Περβάς Πέρες, όπως αντικαθιστά τον κύριο Μπαγιέ. Ναι, εγώ αναπληρώνω τον κύριο Μπαγιέ σήμερα. Θα σας ε, παρουσιάσω τις απόψεις του σε αυτή τη φάση της συζήτησης για τις οικονομικές πολιτικές στην Ευρωζώνη. Ο κύριος Μπαγιέ εκφράζει την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την έκθεση της 14ης Μαρτίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί περιλαμβάνοντας και μια πιο κοινωνική διάσταση στην οικονομική της πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι αφογκράζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο εισηγητής χαίρεται γι' αυτό. Η σύσταση που προτείνει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ε, ε, αντισταθμίζεται από τα κοινωνικά σημεία και την αύξηση των δεξιοτήτων. Επίσης, η σύσταση που αφορά την ε, ενεργό πολιτική στην αγορά εργασίας, οι συστάσεις σχετικές είναι ευπρόσδεκτες γιατί δίνουν ενάψματα για ποιοτικέ ε, θέσεις ε, πλήρους απασχόλησης. Ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες, την κοινωνική αδικία και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποιες συστάσεις για τις ανισότητες των μισθών, για τους φτωχούς εργαζόμενους και την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης. Γι' αυτό και ο εισηγητής ο κ. Μπαγιέ επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Γιατί στο μέτρο που δεν έχουμε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ισότητα και δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, ο κύριος Μπαγκέ θεωρεί ότι θα δυσκολευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι επιθετικοί φορολογικοί σχεδιασμοί για να εξασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση των φορολογουμένων, να διασφαλιστούν τα δημόσια οικονομικά αλλά ταυτόχρονα να έχουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ανισότητες. Επίσης, ε, είναι υπέρ μια φιλόδοξη πολιτικής συνοχής μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών κρατών και περιφερειών. Αυτό είναι θεμελιώδη σημασία για τον εισηγητή. Και από αυτή την άποψη, ο εισηγητή θεωρεί ότι η συνοχή θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και στο μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, γιατί η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική μακροπρόθεσμων επενδύσεων για όλε τι ευρωπαϊκέ περιφέρειες. Στηρίζει την ανάπτυξη και την απασχόληση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και προωθεί καινοτόμε λύσει ε, για τι κλιματικέ αλλαγέ, για την ενεργειακή μετάβαση, την κοινωνική συμπερίληψη αλλά και τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Ο εισηγητής πιστεύει ότι θα καταλήξει σε επικοδομητική συνεργασία με τους συναδέλφους, όπως ε, συνέβη και στην πρώτη φάση αυτού του εξάμεινου εγχειρήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος ε, Τόμ Λάρε είναι ο σκιώδης του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαγιέ για το σχέδιο εκθέσεως, αλλά υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία τα οποία θέλω να θίξω και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα για την ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνη συμφωνούμε ε, στην παράγραφο 26 πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Αυτό δεν πρέπει να υποτιμάται αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η ισορροπία είναι 100% στο κείμενο στην παράγραφο 14 μιλά για τις συστάσεις του Συμβουλίου που θα επιτρέπεται σύμφωνα με αυτή πλεονάσματα να χρησιμοποιούνται για επενδύσεις κλπ αλλά η ίδια σύσταση από το Συμβούλιο λέει ότι θα πρέπει να περιοριστούν οι αμοιβέ. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να τα καλύψω αυτά. Για την παράλογο 16, εκεί γίνεται λόγος για μία μελέτη που συνδέεται με τα πλεονάσματα και τις αυξήσεις των αμοιβών. Θα ήταν καλό να δούμε αυτή τη μελέτη και την στάση που έχει η Ευρωζώνη όσον αφορά το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ζητά κάποιο κάποια πολιτική πιο περιορισμένη. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο εκθέσεως. Θα υποβάλω λοιπόν σχετικές τροπολογίες και άλλες που, τροπολογίες που θα καλύπτουν θέματα του προπολογισμού. Και ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω αφορά την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα, ειδικών για κάθε χώρα. Χρειάζεται να στερνιστούν τα μέτρα αυτά οι χώρες, χρειαζόμαστε άνωθεν προσέγγιση. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες μια άλλη σύσταση αφορά την εφαρμογή των συστάσεων και του σχετισμού των συστάσεων με διάφορες άλλες δομές. Στην παράγραφο 21 ε, αναφέρονται διάφορες εξαιρέσεις. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η αιρεσιμότητα και πρέπει να εφαρμοστεί. Ένα άλλο σημείο αφορά και άλλες συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί. Ε, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πιστεύω ότι δεν καλύπτονται σωστά και αυτά τα θέματα που δεν καλύπτονται σωστά σχετίζονται με, το, με την προσέγγιση συστάσεων αναχώρα και πρέπει από αυτού να εστιαστούμε πριν να ακολουθήσουμε άλλη λύση. Δεν είμαι υπέρ συμπεριλήψεως των στόχων των βιωσίμων, της βιωσίμου ανάπτυξης, διότι εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος να συμπεριλάβουμε πάρα πολλά στο εξάμεινο και το εξάμεινο δεν είχε προβλεφθεί να τα καλύψει όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να γίνει μνήμα ε, στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να καλύπτονται ξεχωριστά. Δεν πρέπει να αναφέρονται εδώ, στα πλαίσια του εξαμήνου. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίλερ δεν μπορούσε να παραστεί και μου ζήτησε να διαβάσω εγώ τη δήλωσή του ο κύριο Ανδαλούς. Θέλει και ο Ζήλερ να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την έκθεσή του. Ο εισηγητής εντοπίζει διάφορα προβλήματα ορθά, με τον ενδεδειγμένο τρόπο και συμμερίζει τι ανησυχίε του εισηγητού για πριν περικοπέ τη πολιτική συνοχή και κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι αντίθετη με το στόχο τη κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ο κ. Ζήλε θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή μα επί του εξή. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούνται από κάποιες χώρες και στην έκθεση επανειλημμένα γίνεται μηνύα σε μέσους όρους και οι μέσοι όροι δεν βοηθούν πάντα ούτως ώστε να διαφωτίζονται οι διαφορές μεταξύ κατών μελών. Γι' αυτό ο κύριος Ζήλα πιστεύει ότι για κάποια ζητήματα η έκθεση θα ήταν καλό να κάνει λεπτομερέστερη περιγραφή. Ο κύριος Ζήλα επίσης σημειώνει ότι ναι μεν γίνεται μηνύα περί των φόρων κάτι που ε, είναι και αρκετά επίμαχο θέμα, αλλά δεν αναφέρεται το θέμα της καλύτερης ίσπραξης φόρων, κάτι που μπορεί να βελτιωθεί σε αρκετά Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που θέλει να τονίσει ο κ. Ζήλε είναι η έκκληση του συγητού για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έχει γίνει ε, θέμα συζητήσεως αυτού και χρειάζεται να υπάρχουν καλύτερα περιθώρια και να υπάρχουν βελτιώσει και εκείνοι που περασπίζονται την ευελιξία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να προσέχουν τι θέλουν. πολύ μεγάλη ευελιξία ίσω να απονομεύσει την όλη ιδέα, όλο το πνεύμα του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Πιο σημαντικό, το τελευταίο Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά αναφέρει ότι τώρα είναι καλή στιγμή για την εφαρμογή των καταλήλων μεταρρυθμίσεων τώρα που πέρασε η κρίση αλλά κάποιοι ακόμα διστάζουν να το κάνουν αυτό, να κάνουν τι αναγκαίε προσαρμογέ μεταρρυθμίσει. Και ο κ. Ζήλε πιστεύει ότι είναι και η ώρα για πολλέ χώρε επιτέλου να κάνουν τη δουλειά του πάνω σε αυτό. Και ο κ. Ζήλε προσβλέπει σε συνεργασία με τον εισηγητή κλπ. κλπ. και να προχωρήσει αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ, Σάντερ, για την άντε. Καρονίλα Χτεκάλ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για το σχέδιο της έκθεσης. Νομίζω ότι αποτελεί καλή βάση συζητήσεων. Πιστεύω ότι θα κινηθούμε και βάσει των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απευθύνει προς τα κράτη-μέλη. Το κύριο στοιχείο των συστάσεων είναι οι εθνικές οικονομίες να ισχυροποιηθούν και εισδήποτε δυσκολίες να μην οδηγούν σε κρίση, να μην οδηγούν άμεσα σε κρίση. Λέμε εμείς στην Ολλανδία ότι καλό είναι να επισκευάσει τη στέγη σου όσο ακόμα υπάρχει λιακάδα, όχι όταν αρχίσουν οι βροχές. Ε, έχουμε πολύ λίγες συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν εφαρμοστεί. Νομίζω ότι η έκθεση κάνει συστάσεις που θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν προσπαθείτε να πετύχετε, να προσελκύσετε επενδύσεις για την κοινωνική πρόνοια, αλλά είναι εσφαλμένη η προσέγγιση. Είναι η προσέγγιση που οδήγησε κατά το παρελθόν σε προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποια, ποιες είναι οι επιτυχείς οικονομίες της Ευρώπης και να δούμε τι κάνουν, να πάρουμε μαθήματα. Οι εταιρείε δίνουν απασχόληση στον κόσμο και όχι οι αρχές. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν θα πρέπει να δαπανά ε, ανεξέλεγκτα ποσά. Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να κάνουν σωστά τις ε, επενδύσεις, να επενδύουν τα χρήματα. οι εταιρείε και οι οικογένειες θα πρέπει να μπορούν να ωφεληθούν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία. Πολλά θέματα προς συζήτηση Προσβλέπω στη συζήτηση και σίγουρα θα καταφέρουμε κάπου να καταλήξουμε σε καλή λύση. Ευχαριστώ Καρολίν. Για τους πρασίνους ο κύριος Ουρτασούν. Ευχαριστώ και εμείς α, ε, ε, θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης είναι καλή βάση για συζήτηση για τις στάσεις χώρα και της πολιτικές ευρωζώνης και μάλιστα μετά τις ε, διακηρύξεις του Μαρτίου έχουμε ε, και τη ε, ε, σχετικά αφήσιμη γερμανική διακήρυξη, τουλάχιστον βλέπουμε ότι ανοίγεται ένας δρόμος για μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, έχουμε αντίφαση αυτής της διακήρυξης σε σχέση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανάγκη μεταρρυθμίσης της Ευρωζώνης. Ε, αυτά τα σημεία θα πρέπει να διευκρινιστούν ε, και να αντικατοπτριστούν στην έκθεση. Ό,τι αφορά τι προτάσει του κ. Μπαγί είναι καλή βάση για τη συζήτηση, αλλά εγώ θα σταθώ σε μερικά σημεία που κρίνω σημαντικά. Συμφωνούμε με το κεφάλαιο για τη φορολογία, ε, δηλαδή να έχουμε φιλόδοξη κοινωνιοποιημένη βάση ε, φορολογίας επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά τις θέσεις απασχόλησης ε, να αναφερθούν οι στάσεις σε ένα χώρα για να εξασφαλίσουμε μια εύρυθμη και δίκαιη αγορά ε, με βάση το κοινωνικό πυλώνα δικαιωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε ανάβασματα για δημόσιες επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα, τις κοινωνικές επιπτώσεις τους. Κάτι που λείπει, κάποια στοιχεία που λείπουν από την έκθεση είναι το ΕΝΤΙΣ, ε, ο προπολογισμό, η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ρόλο ε, τη έκτο δανειστή λύση ε, λύσει έκτακτες περιπτώσει και επίση ανάγκη αυτόματων σταθεροποιητών, όπω είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απασχόληση. Όπως είπαμε, ήδη αρχίζουν ε, και εκπνέουν κάποια προγράμματα νομισματικής πολιτικής, ε, κάτι που μπορεί να υπονομεύσει την ανάκαμψη. Σε ό,τι αφορά τις στάσεις αναχώρα, CSR, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, επικρίνει τα κράτη-μέλη για, για την ενεργειακή του πολιτική που δεν ευθυγραμμίζεται με τις συμπολίες των Παρισίων. Επίσης, ε, δεν φαίνεται από τη στάση αναχώρα μια βελτίωση των ε, συντάξεων. Κρίμα. Επίσης, η διαφθορά εξακολουθεί να είναι μείζο σε πολλά κράτη-μέλη, απειράζοντας αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίση, η στάση αναχώρα θα πρέπει να εγγύψει το ζήτημα τη διαφθορά από ευρωπαϊκή προοπτική. Ε, για, τα ζητήματα, για τα ζητήματα που σα προανέφερα, θα καταθέσουμε τροπολογίε για να βελτιώσουμε το κείμενο. Αποουσιάζει ο κύριος Βιέγκας. Θα ακούσουμε την κυρία Λόπες Βερμέχο. Εμονώ από ευθυντή. Ούτε. Ούτε η κυρία Κάπελ. Δεν ξέρω αν η κυρία Περβάζου Περές θα ήθελε να πει δύο λόγια για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, θα ενημερώσω διεξοδικά τον κύριο Μπαγιέ για το τι υπόθηκε από τους συναδέλφους και νομίζω ότι ε, δεν προδίδω τον εισηγητή να πω ότι η, ο συνδυασμός των ειδικών στάσεων αναχώρα με το ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, είναι αναφυσβήτως γιατί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εξαμήνου υποβάλλονται οι ειδικές συστάσεις αναχώρα. Οι ειδικέ τέσσερα χώρα είναι απόρρια ουσιαστικά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οπότε είναι αλληλένδετα τα θέματα ούτω ή άλλω. Οπότε είναι λογικό να προβληματίζεται ο εισηγητή Μπαγιά για το γενικό πλαίσιο, όπω προσδιορίζεται και λειτουργεί. Σε ό,τι αφορά τη συνδυασμό ε, των στόχων αυτών με τους βιώσιμους στόχους ε, των Ηνωμένων Εθνών ή 21 με τη Συμφωνία COP21, σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό το, του κυρίου Ουρτασούν. Οι ειδικέ συστάσει αναχώρα θα ήθελα να σας πω ότι είναι ένα μέσο εφαρμογής και των ευρωπαϊκών στρατηγικών. Οπότε δύσκολο είναι να θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εφαρμόζουμε τις στρατηγικές αυτές αν δεν παρακολουθούμε το, πεδίο, το επίπεδο εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό προτείνει το σχετικό εδάφιο ο εισηγητής. Τώρα, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη συζήτηση αυτή από τη συζήτηση για τα άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη συζήτηση για το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για παράδειγμα. Και εκεί πιστεύω ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε πλήρως τα δύο θέματα. Και το θέμα του μέλλοντος της πολιτικής συνοχής είναι σημαντικό. Όταν βλέπουμε ε, πώς επηρεάζουν οι δικές ένα χώρα τα θέματα αυτά, δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε μόνο ένα εργαλείο απομονωμένα από τα άλλα. Θα πρέπει να δούμε πώς συνδυάζονται αυτά. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της φορολογίας, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και να βελτιώσουμε την φορησπρακτική ικανότητα των κρατών μελών. Ως προς αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μία αμφισβήτηση του στόχου της ε, μεγαλύτερης ε, φορολογικής εναρμόνισης εκεί που έχει ξεκινήσει. Αυτά γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε πολλές ασχολίες γι' αυτό δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω θα ενημερώσω πάντως διεξοδικά τον εισηγητή. Ευχαριστώ Περβάνος. Η ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 10 Ιουλίου. Θα συζητηθεί το θέμα στις 29 και 30 Αυγούστου. Και θα υπάρξουν ε, ε, συζητήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια στις 19 Οκτωβρίου. Στι 9 μάλλον Οκτωβρίου και στην ΕΚΟΝ θα ψηφιστεί τότε και θα περάσει από την Ολομέλεια στη η του Οκτωβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχουμε κάτι άλλο ε, στα διάφορα υπό το σημείο 8 και υπό το σημείο 9 μπορώ να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι την Δευτέρα 9 Ιουλίου μεταξύ 3 και 6.30 στις Βρυξέλλες αυτό. Και Τετάρτη 11 Ιουλίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 και 9 με 12.30 την 5η 12 Ιουλίου. Να σας θυμίσω ότι απόψε στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προπολογισμών. και θα έρθει εδώ ο Επίτροπος. Καλό σας βράδυ.